Ladies and gentlemen, we are minutes after Επειδή είμαστε 7 λεπτά μετά τις 9 και επειδή οι κύριοι Σκιώδης είναι εδώ, θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Σας καλωσορίζω όλους. Έχουμε δύο κάπως ε, ασυνήθη θέματα, όπου ο εισηγητής και για τα δύο θέματα που θα συζητήσουμε πριν τι ψηφοφορίε ήταν ο κύριο Άντερ Λούνε που έγινε υπουργό ε, άμυνα στην Βελγική Ομοσπονδική Κυβέρνηση. Ο αντικαταστάτη του θα ανακοινωθεί ω Ευρωβουλευτή αύριο. Να τον καλωσορίσουμε στην ΕΚΟΝ. Ω συντονιστή του ECR θα είμαι και πρόεδρο και εισηγήτρια για τα επόμενα δύο θέματα. Συγγνώμη λοιπόν για το θέμα, για το ότι πρέπει εγώ να αναλάβω αυτά τα καθήκοντα. Δεν υπήρχε κανεί ούτε για πρόεδρο ούτε ω εισηγητή. Θα ασχοληθώ και με τα δύο και ελπίζω να ε, μην βαριστείτε να με ακούτε. Το πρώτο θέμα λοιπόν είναι η γνωμοδότησή μα για τη δημιουργία του προγράμματο για την ανταγωνιστικότητα τη ένα αγορά των επιχειρήσεων περιλαμβανομένων των μικρομεσαίων και τι ευρωπαϊκέ στατιστικέ. Ε, Όπω σα είπα, ο κύριο Σάντερ Λούντζ ήταν ο εισηγητή μα. Θα σα διαβάσω λοιπόν το σημείωμα το οποίο μα έχει στείλει. και θα εκπροσωπήσω και τον προηγούμενο και τον εισηγητή που θα τον εγκαταστήσει. Το πλαίσιο πρώτα απ' όλα. Η Επιτροπή μα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τρει τομεί στην πρόταση για το πρόγραμμα τη ενιαία αγορά τι στατιστικέ, την ανταγωνιστικότητα και τι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε. Ιδιαίτερα την εκπαίδευση για τα θέματα Αυτό Ο κύριο Λούνε τονίζει στη γνωμοδότησή του του τρει αυτού τομεί. Πρώτα τονίζει ότι η Eurostat δεν θα πρέπει να είναι θύμα της ε, συγχώνευσης διαφορών προγραμμάτων. Τονίζει τις παραγράφους για τις στατιστικές, χρησιμοποιώντας, χρησιμοποιώντας ε, διευκρινήσεις από το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα. Επίσης, θέλει να ενισχυθεί η κοινοβουλευτική επίβλεψη επί των στρατηγικών και να έχουμε και περιφερειακές στατιστικές όπου είναι δυνατόν. Δεύτερον, για την πολιτική ανταγωνισμού προτείνει να υπάρξουν νέε προκλήσει, να ασχοληθούμε νέε προκλήσει ε, για τα ψηφιακά θέματα και να υπάρξει περισσότερη επίβλεψη για τι δαπάνε των προγραμμάτων τη ενέας αγορά. Και τρίτο και τελευταίο, για τι ε, χρηματοοικονομικές υπηρεσίε, υπενθυμίζει ότι πρέπει να χρηματοδοτήσουμε και μη κερδοσκοπικέ οργανώσει που, που εργάζονται για την κατάρτιση του κοινού για τα θέματα αυτά ε, και να ευνοήσουμε και νέους ετούντες. Έχουμε 88 τροπολογίες από πλευράς των μελών της ΕΛΚ. Θα το αφήσω για λόγους ευγένειας στον εισηγητή να προτείνει ενδεχόμενου συμβιβασμούς. Αλλά τονίζω ότι πολλές από τις τροπολογίες των συναδέλφων υπερβαίνουν ε, τις αποκλειστικές αρμοδιότητες της ΕΚΟΝ και ε, σε περίπτωση αποκλειστικών ε, αρμοδιοτήτων συνήθως υποβάλλεται μόνο μία τροπολογία στην σχετική παράγραφο, άρα έχουμε λιγότερο πεδίο για συμβαστικές τροπολογίες αλλά θα το αφήσω σε αυτόν που σίγουρα θα έχει πολύ κέφι και προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας για τα σημαντικά αυτά θέματα. Αυτά από πλευρά συζητού, οι σκιώδεις λοιπόν για τα σχόλιά τους, για την έκθεση αυτή. Πρώτα απ' όλα για το ΕΛΚ. Η κυρία Τόμεν. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, ως ΕΛΚ στηρίζουμε την πρόταση της Επιτροπής. Είναι καλή. Και θα έχει ως αποτέλεσμα την ε, έγκριση καλών προγραμμάτων για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις μας. Έχω υποβάλει νέα τροπολογίες, τις οποίες θα σας παρουσιάσω αν με επιτρέπετε. Η πρώτη είναι 29, αλλά και η 50. Αυτές οι δύο τροπολογίες θέλουν να τονίσουν το σεβασμό για τους κανόνες ανταγωνισμού. Είναι μια αρχή η οποία ε, ούτως ή άλλως ε, είναι καθιερωμένη στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αλλά καλό είναι να τονίσουμε αυτή την αρχή γιατί έχουν υπάρξει διάφορες περιπτώσεις ε, σε διάφορα κράτη-μέλη όπου δεν έχει γίνει σεβαστή. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι ενισχύσεις του ευρωπαϊκού προπολογισμού δεν ενισχύουν στην ουσία ε, λανθασμένες ε, προσεγγίσεις και ενέργειες. Πρέπει να τονίσουμε τη διεθνή συνεργασία επίσης. Και αυτό είναι θέμα κλειδί για μας. Η εσωτερική αγορά ε, είναι συνεχώς αναπτυσσόμενη, αναπτυσσόμενο εγχείρημα. Στόχος του προγράμματος λοιπόν θα πρέπει να είναι να συμπεριληφθούν και νέες πρωτοβουλίες που όχι μόνο βελτιώνουν την λειτουργία της ενιαίας αγοράς αλλά και αναπτύσσουν περαιτέρω την ενιαία αγορά. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες τροπολογίες που ασχολούνται με την ψηφιακή ενιαία αγορά και εδώ ένα πολύ σημαντικό τμήμα της αγοράς και όλο και αναπτυσσόμενο. Πρέπει λοιπόν να αναπτυχθεί με μεγάλη προσοχή. Είναι ο ε, τάχιστα αναπτυσσόμενος τομέας της οικονομίας μας και αν λοιπόν η νομοθεσία μας δεν συμβαδίζει αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ε, αρνητικά αποτελέσματα, ε, αντίθετα με τις προθέσεις μας. Και επίσης το άρθρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν σε ενωσιακά προγράμματα, ωστόσο έχουν μεγάλες δυσχέρειες. Δεν ενημερώνονται έγκαιρα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα σημείο επαφή. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αναφορά σε ένα δίκτυο που θα μπορούσε να είναι το σημείο επαφή για τι μικρομεσαίε και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ σοσιαλιστές. Ο κύριο Σάντε. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ευρία έκθεση, αλλά νομίζω ότι θα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε. Οι προτεραιότητες για αυτή την πρωτοβουλία, δυστυχώς, δεν έχουν αναφερθεί σωστά. Όσον αφορά τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία, είναι δύσκολο να σχολιάσουμε τώρα οι τροπολογίε 12, 19 και 23 καθορίζουν εκ νέου τον ορισμό των στατιστικών στοιχείων. Παραδείγματο χάρη, το σχέδιο γνωμοτήσεω προσθέτει τη συλλογή των στατιστικών στοιχείων, ενώ εκείνοι που δουλεύουν επί τόπου παρατηρούν τα στατιστικά στοιχεία παράγονται αλλά δεν συλλέγονται και άλλα στοιχεία, ενώ και μόνο δεδομένα και όχι στατιστικά στοιχεία συλλέγονται. Γι' αυτό προτιμώ την αρχική διατύπωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το κείμενο. Πραγματί θα ήθελα να κρατήσουμε την ορολογία που χρησιμοποιείται στον κανονισμό 223 κάθετος 2009 για τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία που αναφέρει σαφώς ότι στατιστικά στοιχεία θα αναπτυχθούν, θα παραχθούν και θα διαβιβαστούν. Περαιτέρω, κάτι χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού δικτύου ανταγωνισμού είναι κάτι άκουσε πρόσδεκτο, κυρίως δοθέντως ότι οι μικρότερες εθνικές αρχές έχουν έλλειψη ανθρωπίνων πόρων και χρημάτων όσον αφορά τη διεξαγωγή θεματικών μελετών. Αυτό ισχύει φαρυπίν όσον αφορά την τροπολογία 6 του εισηγητού. Επίση, υπάρχουν κάποιε τροπολογίε που προτείνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκδίδει εκθέσει για τι εφαρμοστικέ δράσει για την υποστήριξη τη πολιτική ανταγωνισμού για το πρόγραμμα. Επιτροπή Οίκων ίσω να θέλει να προτείνει ένα καλό επίπεδο ελέγχου που θα πρέπει να εξασφαλίσει γύρω στι δραστηριότητε που μετοδοτούνται στο πρόγραμμα ενιαία αγορά και που εμπίπτουν σε αυτή την αρμοδιότητα τη Επιτροπή. Βέβαια, υποστηρίζουμε τη χρηματοδότηση του τομέα των μικρομεσών επιχειρήσεων, κυρίω όταν υπάρχουν συγκεκριμένε επενδύσει ή μικρομεσέ επιχειρήσει που αντιμετωπίζουν φραγμού γεωγραφικής και οικονομικής φύσεω και είναι σε μειονεκτούς περιοχές και τροπολογίε που συμπλεβάνουν αναφέρονται σε ε, κοινωνική επιχειρηματικότητα. Το ενδιαφέρον να εστιαστούμε στη χρηματοδότηση για τον τουρισμό. Όχι συγκεκριμένα αρμοδιότητα τη οίκων, όμως παραμένει ύψη τη σημασία οι διάφορε περιοχέ. Πολλέ επενδύσει στον τομέα απαιτούνται, ούτω ώστε να παραμείνει ανταγωνιστικό τομέα σε όλο τον κόσμο και να αναπτύσσεται με βιώσιμο τρόπο. Η χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να είναι κάτι συνεκτικό με στόχου βιώσιμη ανάπτυξη, όπω καθορίζονται στην θεματολόγιο του ΟΗΕ του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πυλώνα. Άλλη μια προτεραιότητα την ομάδα μου είναι η ενίσχυση τη προστασία των καταναλωτών, των νομικών και οικονομικών του συμφερόντων. Αυτό θα αντικατοπτρίζεται στη θέση του χαρτοφυλακίου μα. Σχετικά με αυτό θα ήταν καλή μια διευκρίνηση τη τροπολογία 21 του σχεδίου γνωμοδοτησίου. Είναι η λογική τη και αναφερθούν αναφορέ στην προστασία των καταναλωτών. Είναι πιθανότατα ότι θα είμαστε αντίθετοι σε αυτό. Τελικά, σε γενική αναφορά, θέλουμε ο πιο αδύνατο κρίκο του εμπορικού κύκλου να μπει πρώτο στι προτεραιότητε του προγράμματο. Γι' αυτό το λόγο υποβάλαμε αρκετέ τροπολογίε που απλώ αλλάζουν την προτεραιότητα και ευνοούμε του πολίτε υπεράνω των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σαντ. Λοιπόν, τρεμόσα από την Άλτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Λούνες, ο οποίος ήταν πολύ αποτελεσματικός και ικανός ευρωβουλευτής και ήταν ευχαριστήσή μας να συνεργαστούμε μαζί του. Και εύχομαι κάθε επιτυχία στον ίδιο και στον αντικαταστάτη του. Αγαπητοί συνάδελφοι, λίγα λόγια θα πω γιατί βεβαίως εμείς οι φιλελευθεροί πάντα είμαστε υπέρ ενό προγράμματος που θέλει να ενισχύσει την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας με ιδιαίτερη αναφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσει Να σας υπενθυμίσω ότι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό επίτευγμα των τελευταίων δεκαετιών είναι η ενιαία αγορά. Αυτό το οποίο μιμούνται σε εμά διάφορες χώρες ανά τον κόσμο είναι αυτές οι ελεύθερες ε, ζώνες κυκλοφορίας ανθρώπων, αγαθών, υπηρεσιών μεταξύ κρατών μελών. Οπότε οποιοδήποτε πρόγραμμα της Κομισιόν για να βελτιώσει την ενιαία αγορά ε, είναι προς ε, το συμφέρον μας. Και επίσης βλέπουμε πάρα πολύ θετικά το ότι υπάρχει μια ειδική αναφορά για τις μικρόμεσες επιχειρήσεις. Όπως ίσως ξέρετε, ναι, και οι πολυεθνικές είναι πάρα πολύ σημαντικές εταιρείε, αλλά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνεισφέρουν κατά κύριο λόγο στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εγώ είμαι από την Βαρκελόνη, η χώρα μου, η Καταλωνία, έχει 8.000 πολυεθνικές, αλλά 500.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις δημιουργούν 90% των νέων θέσεων εργασίας. Γι' αυτό χαιρόμαστε το ότι η Κομισιόν ε, θεωρεί απαραίτητο να αυξήσει τα εργαλεία ενημέρωσης και εκπαίδευσης ε, και μηχανισμούς ε, εκτάκτου ανάγκης για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό το ότι αυτό αφορά τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία γιατί πρέπει να έχουν αυτοί οι οποίοι χαράζουν πολιτική τις ε, καλύτερες πληροφορίες και τα μέσα για την διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι' αυτό ακριβώ χαιρόμαστε για το ότι τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία αποτελούν επίσης έναν στόχο της Κομισιόν προς βελτίωση, εναρμόνιση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών. για την βελτίωση της ποιότητας ε, των στατιστικών στοιχείων και γι' αυτό, αυτό ακριβώς ε, θέλουμε να βρούμε ένα συμβιβασμό με όλες τις ομάδες ε, για το θέμα αυτό. Και τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε διαφορετικά κρατημέλη υπάρχουν περιφερειακά κοινοβουλία με προϋπολογισμό δικό τους και μια μεγάλη παράδοση που έχουν πολύ καλές στατιστικές υπηρεσίες και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Οπότε είμαι στην διάθεσή σας για την συνεργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιο εδώ εξ των Πρασίνων. Όχι. Από την ΚΟΕ. Κάποιος άλλος θέλει τον λόγο. Όχι τότε ως συζηγήτρια θα συνοψίσω εγώ να ευχαριστήσω τους και συζητητέ για όλα τους ε, τα σχόλια τα οποία σημείωσα εδώ θα φροντίσω ε, νέος συζηγητής να τα έχει και είμαι σίγουρος ότι και το προσωπικό θα φροντίσει για την ενημέρωσή του. Το χρονοδιάγραμμα είναι το εξή. Σοφορία στην Επιτροπή είναι 10 Δεκεμβρίου, οπότε σας ε, ζητώ να συνεργαστείτε με τον νέο συνάδελφο που θα έρθει αύριο για να περάσει αυτό το θέμα στην ώρα του στις 10 Δεκεμβρίου. Αυτά σας ευχαριστώ. Τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Περνάμε στο επόμενο. Λοιπόν, για μια ακόμη φορά το επόμενο σημείο. Διατάξεις διευκολύνει τη χρήση οικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και τη δίωξη ορισμένων ποινικών δικημάτων. Ο νέος ηγετής, ο Μπεντ Λούκε, δεν είναι εδώ, οπότε εκ νέου θα τον αντικαταστήσω ως εισηγητή και θα διαβάσω τις σημειώσεις που μου έδωσε. Ο κ. Λουκ ζητά συγγνώμη που δεν παρίσταται και δεν συμμετέχει στη συνεδρίαση. Μου ζήτησε να διαβάσω το εξή κείμενο εκ μέρου του. Ο κ. Λούκη ευχαριστεί τους σκιώδει εισηγητέ και τον προκάτοχό του, τον εισηγητή, τον κ. Σαντολούνε, για την έξοχη και επικοδομητική εργασία του. Όλοι οι συνάδελφοι έχουν κοινό στόχο, διευκόλυνση την ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν την καταπολέμηση του ξεπλήματο χρήματο και τη χρηματοδότηση των νομοκρατών μεταξύ εθνικών μονάδων, ερευνήσεω οικονομικών θεμάτων και άλλων αρχών, ταυτόχρονα προστατεύονται τα θεμετά συμφέροντα φυσικών νομικών προσώπων, ενδεχομένω θα μπορούσαν να επηρεάζονται από τι πληροφορίε. Πετύχαμε συνένεση στα περισσότερα σημεία με μόνο μικροδιαφορέ απόψεων που απομένουν. Και ο Λούκη ελπίζει ότι η γνωμοδότηση θα τύχει ευρεία υποστηρίξεω στην Επιτροπή Οίκων και ελπίζουμε να πετύχουμε του στόχου ε, του συμπεφωνημένου. Αυτό είναι το τέλο των σχολείων του Σιγητού. και θα ήθελα να καλέσω τους σκιώδεις να σχολιάσουν για το ΕΛΚ ο κ. Βαντεκαντελάμπε, Καντελάερ, που δεν είναι εδώ, κάποιος άλλος εκ μέρου του ΕΛΚ που θα ήθελε να λάβει το λόγο και να μιλήσει στη θέση του, εν τη αυτή η περίπτωση, ο κ. Σκόφορντ από τους σοσιαλιστές. Κάποιος από τους σοσιαλιστές που θα ήθελε να μιλήσει εκ μέρους της ομάδας. Ορίστε. Ο Σκιώδης, ο κύριος Κόφορντ, θα ήθελε να ευχαριστήσει τον εισηγητή και εκ μέρου ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα ήθελε να προβεί σε κάποια σχόλια. Χαιρόμεθα που ευρέθησαν συμβιβαστικές που μπορούν να λειτουργήσουν για το μεγαλύτερο κομμάτι του ε, κειμένου και έχει ενισχυθεί εν σχέση με την αρχική εκδοχή του κείμενου, σημαντικά. Συμβάλαμε με αρκετέ τροπολογίε και εμεί και χαίρεται που βλέπει ότι οι περισσότερες από αυτέ αντικατοπτρίζουν το κείμενο. Εξασφάλιση αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ 100 μελών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και των σχετικών αρχών για την ε, διερεύνηση, εξυχνίαση, δίωξη, ε, πρόληψη, εντοπισμό και τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων είναι ύψιστη προτεραιότητα για την ομάδα μα, μια προτεραιότητα που βεβαίως συνδέεται στενά με, τα, με τις προσπάθειες που καταβάλλουν σε αυτή την ε, Επιτροπή και στην Επιτροπή ε, Tax 3 και κάνουμε άλλο ένα βήμα εδώ για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας κατά του οικονομικού εγκλήματος, όπως είναι τα θέματα του ξεπλήματος χρήματος. Είναι ένα βήμα που σαφώς απαιτείται μετά την πρόσφατη σειρά σκανδάλων ε, νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων που διαπιστώθηκε σε διάφορες ε, ευρωπαϊκές τράπεζες γνωρίζουμε ότι σε αρκετέ περιπτώσεις η, μία, η αναποτελεσματική συνεργασία μεταξύ αρμοδίων φορέων έχει καθυστερήσει, παρεμποδίσει και τον τοπισμό και την εξυχνίαση αυτών των ε, αδικημάτων και θέλουμε ταχεία έγκριση και εφαρμογή των νέων ε, ενισχυμένων διατάξεων για την ταχύτερη ανταλλαγή ζωτικής σημασίας πληροφοριών που σχετίζονται με ποινικά δικήματα και αν επιτρέπετε να προσθέσω σε αυτά που αναφέρθηκαν από το σκιώδη συγκητή θα ήθελα να πω ότι για μας είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη θητεία να μην αποδυναμώσουμε κανένα από τα επιτεύγματα που έχουν υλοποιηθεί εντός αυτής της Επιτροπής όταν υθετήσαμε την, το προηγούμενο νομοθεσία ε, και συνεχίζονται συζητήσεις σχετικές και σε άλλες επιτροπές όπου ξέρουμε ότι διάφορες εθνικέ μονάδες εξυχνίασης οικονομικών εγκλημάτων έχουν καλό ιστορικό παρελθόν, αλλά αυτός δεν είναι λόγος να μην βελτιωθεί το πνεύμα συνεργασίας. Θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών των διαφόρων κατών μελών. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλου κοιόδη. Κάποιο άλλο εκπρόσωπο άλλη πολιτική ομάδα που θα να τοποθετηθεί. Εν τε αυτή περιπτώση ολοκληρώνεται αυτό το τμήμα της συνεδριάσεως για τη συζήτηση επιτροπολογιών. Επενθυμίσω, η ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ είναι σήμερα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ολοκληρώνεται αυτό το τμήμα της συνεδριάσεως. Ένα διάλειμμα πέντε λεπτών μέχρι ότου ξεκινήσει η ψηφοφορία μας. Ευχαριστώ πολύ.

Ωραία, λοιπόν, ε, βλέπω ότι είμαστε κάπως περισσότεροι, οπότε μπορούμε να αρχίσουμε τις ψηφοφορίες. Είναι σύντομες. Δεν θα πάρουμε πολύ χρόνο, ελπίζω. Λοιπόν, καταρχάς, ε, θέλω ξεκινώντας να ευχηθώ στον δόκτωρα Λάγεν χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του. Λοιπόν, ε, είναι πολύ καλή ευκαιρία για να κάνουμε και μια ψηφοφορία ελέγχου, μια δοκιμαστική ψηφοφορία παρακαλώ. Ε, συνάδελφοι, πριν ψηφίζουμε να ε, αναφέρω ότι ανησυχώ ιδιαίτερα ότι το κοινοβούλιο μας μοιάζει να είναι έτοιμο να αποδεχθεί μια πρόταση για το CNS που αλλάζει την κατάσταση με βάση το άρθρο 121.6 ε, όχι μόνο για τους μεσοπρόθεσμους στόχους αλλά και άλλους κανόνες όσον αφορά τα δημοσιονομικά, τα χρηματοπιστωτικά μάλλον. Και μάλιστα αυτό γίνεται με άλλη νομική βάση. Το 126.14 αυτό στην πράξη θα σημαίνει ότι αποδεχόμεθα ότι κάτι το οποίο έχουμε ψηφίσει μέσω συναπόφαση θα γίνει τώρα απλή διαβούλευση με γνωμοδότηση. Εάν το Κοινοβούλιο αποδεχθεί αυτή την περιορισμένη νομική βάση, εγώ θα προσφύγω στο δικαστήριο κατά του Κοινοβουλίου, διότι παραβιάζει τα δικαιώματά μας όλων ημών ως ε, Ευρωβουλευτών που δικαιούμεθα στην απόφαση με βάση τις συνθήκες. Λοιπόν, θα, το, θα κάνουμε τα δέοντα λοιπόν και η Γραμματεία και η Προεδρία. Αντί αυτή περιπτώσει περιπτώση, ξεκινήσουμε με δοκιμαστική ψηφοφορία. Παρακαλώ, χρησιμοποιήστε τις κάρτες σας και ψηφίστε. Θα κάνουμε τη δοκιμή. Δύο κάρτες λείπουν. Κύριε Κόνι, δεν έχετε κάρτα, έτσι. Ωραία. Θα προσπαθήσουμε να προσθέτουμε κάθε φορά την ψήφο σας όταν αυτό έχει κρίσιμη σημασία. Λείπει ε, μία ψήφος εν συγκρίση με τον αριθμό των καρτών που εισήχθησαν. Όλοι οι παρόντες, όλοι ξέρετε πώς χρησιμοποιείτε τις κάρτες σας. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν την πρώτη ψηφοφορία αφορά το σχέδιο νομοθετικής εκθέσεως Giggold για το πρόγραμμα φυσικάλης για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογήσεως. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Παρακαλώ, υπομονή είναι η πρώτη ψηφοφορία μου ως Προέδρου. Όποιος ξέρει, με ξέρει, ξέρει, δεν ξέρω πολύ καλά πώς να μετρά από αυτή τη θέση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Okay, so the vote is rejected. Απορρίπτεται 19-16. Τροπολογία 9 απεσύρθη. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική α υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 74 υπέρ. Κατά Αποχές έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 24-21 συμβαστική β υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική C υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται συμβαστική D τρεις προφορικές τροπολογίες έχουμε εδώ υπάρχουν αντιρρήσεις σχετικά με τις προφορικές τροπολογίες αντί αυτή την περιπτώση υπέρ πρώτης τροπολογίας κατά άποχες προφορικές τροπολογίες εγκρίνονται Δεύτερη τροπολογία, υπέρ. Κατά. Άποχες. Θα πρέπει να γίνει έλεγχος. Έλεγχος για τη δεύτερη προφορική τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτη προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος φοβάμαι άρχεται πέρα ψηφοφορίας με μεγάλη διαφορά εγκρίνεται δεν ξέρω πως δεν το είδα πάμε στο επόμενο σημείο Η γραμματεία λέει αν θέλετε να ψηφίσουμε τη συμβαστική στο σύνολό τη, μπορούμε να το κάνουμε υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική ε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική FA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Budget 13 υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. 109 budget υπέρ, κατά, αποχές, ξανά έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, απορρίπτωται. 110 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 112. Με προφορική τροπολογία των πρασίνων. Υπάρχουν αντιρρήσει την προφορική τροπολογία. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ήττα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Εγκρίνεται διορθώνει η Πρόεδρος. Ζητώ συγγνώμη. 44 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται συμβαστική IA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται συμβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική και υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική μη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 64 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, εγκρίνεται, 65 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε η μονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Σαφώς εγκρίνεται, οπότε το θέμα θα προθεθεί στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Δεύτερη ψηφοφορία. πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για διατάξεις ε, για δημοσιονομική υπευθυνότητα στους μεσοπρόθεσμου προπολογισμού των κρατών μελών. Τροπολογίες 8, 9, 10, 11, 12 μαζί, υπέρ. Να ζητώ συγγνώμη με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχια τη ψηφοφορία. Πέρας. Αχα. Απορρίπτεται. λένε εδώ ότι είναι τροπολογία η οποία απορρίφθηκε, οπότε συνεχίζουμε με τον υπόλοιπο κατάλογο ψηφοφορίας. Λοιπόν, συμβαστική α υπέρ, κατά, αποχές, ε, θα πρέπει να το επαληθεύσουμε, αρχή ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική βήτα υπέρ. Ε, ζητώ συγγνώμη. Τροπολογία 39 έχει καταπέσει. Ε, μάλλον τροπολογία 39 υπέρ. Κατά. Αποχές θα πρέπει να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία πέρας. Εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να την παληθεύσουμε άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική β' υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται άρθρο 2 42 υπέρ Υπάρχει έτοιμα για χωριστή ψηφοφορία στην 42 υπέρ κατά αποχές πρέπει να την επαληθεύσουμε αρκετή ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται συμβαστική γάμα υπέρ κατά αποχές Πρέπει να την επαληθεύσουμε κάτι γίνεται εδώ πέρα με τα νούμερα. έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Πρέπει να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ε, κάντε λίγο υπομονή γιατί είναι τσίμα τσίμα οι ψηφοφορίες. Λοιπόν, 47 υπέρ. Κατά αποχές να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρας απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές πρέπει να την επαληθεύσουμε και αυτή να έρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 49 υπέρ Κατά. Πρέπει να τα παληθεύσουμε και αυτήν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Η ισοψηφία άρα απορρίπτεται. 50 υπέρ κατά αποχές πρέπει να την επαληθεύσουμε και αυτήν. Οι μεγάλες ομάδες δεν είναι πια προβλέψιμες, λοιπόν άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τι υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε αρχιετή ψηφοφορία πέρας απόρριπτεται 55 υπέρ κατά αποχές να την επαλτεύσουμε Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική η υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές πρέπει να την επαληθεύσουμε αρκετή ψηφοφορία. Πέρας. απορρίψετε 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές πάτε να παληθεύσουμε αρχιτή η ψηφοφορία πέρας η ισοψηφία άρα απορρίπτεται έχουμε την 60 τώρα υπέρ κατά αποχές πρέπει να επαληθευτεί έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Η ισοψηφία άρα απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά αποχές. Πρέπει και αυτή να επαληθευτεί. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 62 υπέρ κατά αποχές πρέπει να την επαληθεύσουμε ε, υπομονή παρακαλώ θα τις ε, κοιτάμε τις περισσότερες γιατί άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 63 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε. Α, έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65 υπέρ. 64 τέσσερα λοιπόν να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 65 πέρα. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την επαληθεύσουμε αρκετή ψηφοφορία. Πέρας. Απόλυπτεται 65 υπέρ. Δεν σηκώνει κανείς το χέρι, δεν ξέρω τι γίνεται. Ε, Φτάνει που είναι τόσο δύσκολο, αλλά ε, άμα δυσκόνται και το χέρι. Υπάρχουν αντιρρήσεις να γίνουν όλες ηλεκτρονικά, γιατί είναι πολύ κοντά τα αποτελέσματα. Λοιπόν, θα γίνουν όλες ηλεκτρονικά. Η 65 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 66. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. G. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Η ισοψηφία και απορρίπτεται. Τροπολογία 5 λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Ισοψηφία απορρίπτεται. 67. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική H με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 72 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρας δεκτή 77 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 78 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 79 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 80 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 81 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Απορρίπτεται. 82. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 83. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απόρριπτε. 85 άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας. το 86 άρχιτε ψηφοφορία. περα Απόρριπτε. Συμβαστική I υπέρ... Ε, ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. 87. Άρχεται τη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. 88. Άρχεται τη ψηφοφορία. Πέρας. το J. Ηλεκτρονική ψηφοφορία και πάλι άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε με μία ψήφο διαφορά. Οπότε ψηφίζουμε την ε, 14 σε δύο μέρη μέρος πρώτο άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορριφθήκε μία ψηφοφορία φορά. Συμβαστική κάπα, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. L, συμβαστική άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Να απορριφθείτε. Απολογία 16 άρχεται η ψηφοφορία. πέρας απορρίπτεται 17 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται συμβαστική M άρχεται η ψηφοφορία πέρας Ισοψηφία απορρίπτεται. Λοιπόν, ψηφίζουμε 18, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 19, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική νη. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε λοιπόν στις τροπολογίες. 20. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 21 άρχεται ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται η τροπολογία 22 άρχεται ψηφοφορία πέρας 23 άρχεται ψηφοφορία Πέρας. Απορρίπτεται. Η 24. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Να απορρίπτεται η 25. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Να απορρίπτεται η 26. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 27, αρχιτή ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 28 αρχιτή ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 29 αρχιτή ψηφοφορία. πέρας η ισοψηφία και απορρίπτεται 30 άρχεται η ψηφοφορία πέρας και πάλι απορρίπτεται 31 με ηλεκτρονική ψηφοφορία Πέρας. Απορρίπτεται. 32 αρχιτή ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική όμικρον άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Οπότε περνάμε στις τροπολογίες. 34, αρχιετή ψηφοφορία. Πέρας. Κατέπεσε η συμβαστική, πρέπει να κάνουν τροπολογίες, είναι δύο στη συγκεκριμένη συμβαστική. χωριστές ε, στην 34, ε, 35 και 33. Χαίρομαι που δεν υπάρχει διαδικαστικό πρόβλημα, οπότε ψηφίζουμε την 33, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 34, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 35, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική πι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 36 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 37 αρχή ψηφοφορία. Πέρας. Απόλυπτεται 38 αρχή ψηφοφορία. Πέρας. Ε, εγκρίνεται. Να ρωτήσω τον εισηγητή αν έχει αποσυρθεί η προφορική τροπολογία. Ωραία. Τότε περνάμε στο εκτιμώντας 1, τροπολογία 13, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ναι, είναι ονομαστική ψηφοφορία στο κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ισοψηφία, άρα απορρίπτεται. Λοιπόν, λοιπόν, η Επιτροπή μας δεν ενέκρινε την έκθεση στην ε, μορφή που έχει τώρα. Τρίτη μας ψηφοφορία. κυρία Χρύπνερ. Οπότε η επιλογή που μας μένει είναι η πρόταση της Επιτροπής. Νομίζω ότι θα πρέπει να ε, ενημερωθούμε για το πώς έχουν τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο περιπλοκή η κατάσταση. Δεν θα σας πούμε με βάση τις απόψεις που εκφράζονται εδώ στο Προεδρείο. Θα ε, ζητήσουμε ε, να μας δοθούν ε, να, μας δοθεί, να μας δοθούν συμβουλές για το τι σημαίνει το γεγονός ότι εμεί απορρίψαμε αυτή την έκθεση σε σχέση με την πρόταση επιτροπής. Λοιπόν, τρίτη ψηφοφορία σήμερα το πρωί για το σύστημα μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρησης για τις παραδόσεις αγαθών. Η πρώτη ψηφοφορία ονομαστική άρχεται. Περιμένετε να ψηφίσετε, περιμένω να ψηφίσετε όλοι. Όσο, όσο, αν ναι, τα πάτε πιο γρήγορα, προλαβαίνουμε. Πέρας. Απολύτω. Τροπολογία 30. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 5. Α, όχι. Εφόσον ενεκρίθη η 30 πρέπει να περάσουμε στη 32. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 6 καταπίπτει 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 8. <clears throat> Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή 12 υπέρ. Α, συγγνώμη, ήταν ταυτόσιμες, οπότε έπρεπε να έχουν ψηφιστεί μαζί. 13 λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την ελέγξουμε. Πέρας. απορρίπτεται κατηγορηματικά, αλλά σας παρακαλώ ε, δεν σηκώνετε τα χέρια σας με τον αντίστοιχο τρόπο. Δεν έβλεπα εγώ τόσο κατηγορηματική απόρριψη. 37 παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, συγγνώμη, απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 38 υπέρ κατά αποχές δεκτή όχι απορρίπτεται ε, τουλάχιστον οι δύο συντονιστέ να μου λέτε τι γίνεται, γιατί δεν καταλαβαίνω. Απορρίπτεται λοιπόν. 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή 41 καταπίπτει 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή 21 υπέρ κατά αποχές Δεκτή. Τροπολογία 1 στην αιτιολογική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 25 κατά πίπτη, 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 26 κατά πίπτη, 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ψηφίζουμε τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής σε ονομαστική ψηφοφορία άρχεται πέρασε 24 υπέρ, 7 κατά, 16 αποχές, εγκρίνεται. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Επόμενη ψηφοφορία. Για την νομοποίηση προϊόντος εγκλήματος. Συμβαστική α υπέρ, κατά αποχές, δεκτή. 8 υπέρ, κατά αποχές, να ελέγξουμε. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Με δύο ψήφους διαφορά. Αν συμφωνείτε, επειδή ε, είναι η ίδια παράξενη, ο ίδιος παράξενος σχεσμός, να να κάνουμε πάντα ονομαστικές ψηφοφορίες. Τροπολογία 9. Άρχεται. Πέρας. Εδώ δεν χρειαζόταν βέβαια ηλεκτρονικό έλεγχο. Εν να επιχειρήσουμε και πάλι δια ανατάσσεω 10 υπέρ κατά αποχέ δεκτή. 11 υπέρ κατά αποχέ. Τώρα χρειάζεται έλεγχο. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 45 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 12 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 13 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 46 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 47 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 14 υπέρ. Κατά Αποχές δεκτή. 48 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 49 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 50. Α, έχει αποσυρθεί. Συμβαστική B υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική C υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές δεκτή 57 υπέρ κατά αποχέ, ε, αποχές δεκτή 58 υπέρ κατά ε, αποχές απορρίπτεται συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές δεκτή 60 υπέρ κατά αποχές δεκτή 61 υπέρ κατά αποχές δεκτή 62 υπέρ κατά αποχές δεκτή 17 κατά πίπτη 63 63 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 64. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές παλήθευση για τη 19 άρχεται πέρας ψηφοφόρια. εγκρίνεται συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση ηλεκτρονική ξεκινάει τώρα πέρας εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ξεκινάει η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική ήτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική γιώτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση άρχεται πέρας εγκρίνεται ψηφίζουμε τι Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο τροποποιήθη η ονομαστική ψηφοφορία άρχεται πέρας 43 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος εναντίον και δύο αποχές. Οπότε εγκρίνεται από την Επιτροπή. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Επόμενη ψηφοφορία. Σχέδιο εκθέσεως και ανταμάτω. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την ετήσια έκθεση αυτής. Πρώτη ψηφοφορία. Τροπολογία 55 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται σημαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Σ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική DA ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 91 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 92 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 94 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος άρχεται πέρας απορρίπτεται τροπολογία 95 υπέρ φαίνεται ότι καλύπτεται 95 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τοπολογία 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η επόμενη καλύπτεται 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 118 υπέρ Ακαλύπτεται 118. Συμβαστική F υπέρ. κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Ήτα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται ένα υπέρ κατά αποχές επαλήθευση ηλεκτρονική ξεκινάει τώρα τέλος απορρίπτεται 142 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση άρχεται Πέρας. Απορρίπτεται. 143. Το αρχικό κείμενο πρέπει να ψηφίσουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική γιώτα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Comp ε, Sustainability. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική J, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική K, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 167, καλύπτεται. Συμβιβαστική. Συμβαστική επί της παραγράφου 13 μου κάνετε τη ζωή μου δύσκολη. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική L. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, Εγκρίνεται. 175 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 176 καλύπτεται. 177 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 178 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση για την 178 ξεκινάει τώρα πέρας απορρίπτεται 179 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική μη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 183 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θα κάνουμε έναν έλεγχο ξεκινάει βλέπω ότι εγκρίνεται μεγάλη διαφορά τέλος πάνω πέρας 30 ψήφοι υπέρ 184 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτονται. 186 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτονται. 187 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 188 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτονται. 189 υπέρ κατά αποχές έλεγχος παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 190 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 192 το αρχικό κείμενο παράγραφος 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 192 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 192 άρχεται η ψηφοφόρια. Δεν ήταν ξεκάθαρο με τόντας χέρια. Πέρας. Απορρίπτεται. 193. Υπέρ. Κατά. Πρέπει να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική νη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 197 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 201 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική όμικρον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική P υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 226 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 227 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 214 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται θα γίνει έλεγχος για τη 214 άρχεται πέρας απορρίπτεται 216 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική R υπέρ με προφορική τροπολογία, νομίζω. Υπάρχουν αντιλήσει την προφορική τροπολογία. Δύο προφορικές τροπολογίες. Πρέπει να ψηφίσουμε τις δύο προφορικές τροπολογίες ξεχωριστά. Πρώτη προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές, έλεγχος, άρχια τη ψηφοφορία για την πρώτη προφορική τροπολογία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η δεύτερη. Προφορική τροπολογία υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συνεπώς. Ψηφίζουμε όλο το κείμενο, όλη τη συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται συμβιβαστική. Δεν βλέπω τα χέρια του ΕΛΚ. Κάποιος μπορεί να αντικαταστήσει. 228. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το αρχικό κείμενο. Παράγραφος 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 230 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος ξεκινάει. Πέρας. Μετακινήθηκαν τα χέρια, παρακαλώ, να είναι ξεκάθαρη η ψήφος. Να μου κάνει τη χάτη, σηκώντε το χέρι. Τροπολογία 1 της συντηλογής αναφοράς 1, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται τρία υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται πέρας εγκρίνεται το 4 υπέρ κατά αποχές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 αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αρχικό κείμενο τελική αναφορά 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 21 υπέρ κατά, υπέρ μάλλον συγγνώμη, κατά, αποχές εγκρίνεται, 22 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 23 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Σημαστική S υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 27 υπέρ, Δεν βλέπω τα χέρια της Άλντε υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία για την 27. Πέρας. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Σημαστική ταφ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Σημαστική γιου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική W υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Χ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική Y υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Ζ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές και πρέπει να γίνει έλεγχος που ξεκινάει τώρα πέρας εγκρίνεται ονομαστική ψηφοφορία για το τροποποιημένο κείμενο ξεκινάει Πέρας. Εγκρίνεται. 39 ψήφοι, 2 ψήφοι κατά, 3 αποχές. Ευχαριστούμε γιατί. Τελική ψηφοφορία που έχουμε σήμερα το πρωί. Σχέδιο εκθέσεις πρωτοβουλίας Τόλβαλτς για την Τραπεζική Ένωση και τη σχετική της έκθεση. Συμβαστική Α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική γάμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 92 υπέρ κατά Θα έπρεπε να την επαληθεύσουμε αρκετή ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική J υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική K υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1-1-5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 118 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε αρχιετή ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται σημαστική εν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ομικρόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πι, υπέρ κατά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 143 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 153 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε αρχή της ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται συμβαστική RA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 152 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστικές υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 163 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 168 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 171 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε άρχεται Προφανώς απορρίπτεται τώρα εδώ που το βλέπω. 170 ε, υπέρ κατά εποχές δεκτή. Αρχικό κείμενο της παραγράφου 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 172 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συνεργαστική γιου υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 183 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 184 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 185 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 186 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Αρχικό κείμενο της αιτιολογικής αναφοράς 1 θα τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Αιτιολογικές αναφορές 1, 2, 3 και 4 υπέρ. Κατά αποχές δεκτές. Αιτιολογική αναφορά 5, τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά αποχές γκρίνεται. Αιτιολογική αναφορά 6, αρχικό κείμενο και 7 μαζί υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. αποχέ, Δεκτή. Αιτιολογική αναφορά. 8. Τροπολογία 4. Αρχικό κείμενο. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Αιτιολογική αναφορά 8α4. Ε, ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή αρχικό κείμενο για τις 9 έως 11 μπλοκ υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ 6 έως 10 όλες μαζί υπέρ κατά αποχές δεκτή εκτιμώντας τροπολογία 11 έχουμε μια τροπολογία 10 6, 2, 10 ήταν λοιπόν εκτιμώντας τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή 16 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Ναι, απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο. Δεκαοχτώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. εννέα υπέρ. Κατά. Αποχές πρέπει να το επαληθεύσουμε αρχή τη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές να τα παληθεύσουμε. Αρχιετή ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Αρχικό κείμενο. Δεν ναι, το ψηφίζουμε. 26 υπέρ, κατά, αποχές απορριφθεται 27 υπέρ κατά αποχές απορριφθεται αρχικό κείμενο λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές πρέπει να την επαληθεύσω Αρχιετή ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές πρέπει να επαληθευτεί αρχή η ψηφοφορία πέρας δεκτή 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή 29 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε πέρας δεκτή 30 καταπίπτει 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε Πέρας απορρίπτεται 35 υπέρ. Κατά. Με Αποχές. Πρέπει να την επαληθεύσουμε αρκετή ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την πρόταση κομισιόν όπως τροποποιήθηκε. Ζητώ συγγνώμη. Ε, εδώ πέρα μου διαβάζουν ότι μου έχουν γράψει. Όχι αυτά που πρέπει να πω. Αποτυχημένη πρόεδρος, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, τίθεται σε ονομαστική ψηφοφορία. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Δύο ακόμη πρέπει να ψηφίσουν, μεταξύ των οποίων και εγώ. Πέρας. Δεκτή. 35 υπέρ, 5 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια στον συγητή. Τώρα διακόπτουμε για 5 λεπτά πριν την κοινή συνεδρίαση στις 11 η ώρα. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Bye.